συζήτηση έκθεση του συναδέλφου κ. Γιάννος Όντερ με τίτλο «Έλεγχος των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες». Θέση εισηγητή, καταλαμβάνει, θέση εισηγητού καταλαμβάνει ο συνάδελφος κ. Ρίχαρτ Ζέιμπα και έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκπροσωπώ εδώ τον πρώην συνάδελφο Γιάννο Σάντερ ο οποίος διεκπέρασε αυτή την έκθεση. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω και να του ευχηθώ καλή τύχη. Όπως γνωρίζετε ανέλαβε πρόεδρος της Δημοκρατίας στην Ουγγαρία και είναι πολύ σημαντικό να έχει η Ουγγαρία ένα τέτοιο πρόεδρο, ε, κάποιον που έχει τόση στενή επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Περί πρόκειται στην παρούσα οδηγία. Πρόκειται για μια προσαρμογή ε, της οδηγίας σε Βέζο 2. Πρόκειται κυρίως για την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων με ε, χημικές ουσίες όπως έγινε στο Σεβέζο, Σφάιτσαρ, Χάλη στην Ελβετία και αλλού ή όταν συμβούν να έχουμε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για το περιβάλλον και για τους ε, πολίτες. Νομίζω ότι η Σεβέζο 2 ε, ήταν μια οδηγία που πέτυχε αρκετά, τώρα καλούμαστε να την προσαρμόσουμε διότι ακριβώς αυτή η οδηγία ε, αφορά την επισήμαση συσκευασία ε, αλλά και ταξινόμηση αυτών των ουσιών, η λεγόμενη οδηγία CLP και την 1η ε, Ιουνίου 2015 τίθεται σε ισχύ. Εξού και το παράρτημα 1 της οδηγίας ΕΒΕΖΟ 2 που απαριθμούνται επικίνδυνες ουσίες και είναι το πεδίο εφαρμογή για τις εταιρείε. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η προσαρμογή. Στην Ευρώπη έχουμε περίπου 10.000 χημικές εταιρείε που θίγονται άμεσα γιατί παράγουν ε, τέτοιε ουσίε και θα ήθελα να προσθέσω εδώ και είναι σημαντικό ιδιαίτερα στην Ευρώπη είναι μεγάλη η χημική βιομηχανία και θα πρέπει να τη διατηρήσουμε. Προηγουμένω συζητήσαμε για τη θέση απασχόληση και χρειαζόμαστε αυτή τη βιομηχανική βάση για να εξασφαλίσουμε στο διηνικές ε, τι θέσει. Θα πρέπει όμω να εξασφαλίσουμε ταυτόχρονα να προστατεύονται οι άνθρωποι όπω και το περιβάλλον από κινδύνου που απορρέουν από τέτοια εργοστάσια να αυξηθεί η προστασία θέλουμε, όχι να μειωθεί. Εκεί στοχεύει η αναπροσαρμογή και θα πρέπει να ποντάρουμε ακριβώς εκεί και στην καλύτερη εφαρμογή αλλά και στις ίσους ε, όρους και κανόνες ε, ανταγωνισμού μεταξύ των εταιριών προσπαθήσαμε να προσαρμόσουμε και γενικά, δηλαδή ε, η διοικητική επιβάρυνση να είναι όσο γίνεται μικρότερη σε όλη την Ευρώπη είναι μεγάλη πρόκληση και δυσκολία για εμάς τους Ευρωπαίους γιατί πολλοί ανταγωνιστές μας στον κόσμο έχουν πάρα πολύ χαλαρές ε, ρυθμίσεις ε, και πλήττονται πολλοί δικές μας εταιρείε από αυτό. Άλλος λόγος για την προσαρμογή επίσης ήταν και η Σύμβαση Άρχους. Γνωρίζουμε ότι αυτή είναι μια σύμβαση που έχει υπογραφεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για καλύτερη ενημέρωση του κοινού και πρόσφαση ε, στο δικαστικό σύστημα και αυτό έχουμε τώρα ε, επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις και ο κόσμος που ε, ζει και μένει πολύ κοντά σε αυτές τις επιχειρήσει να έχει και αυξημένη πληροφόρηση και δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη. Τα βασικά προβλήματα θα είχαμε το Συμβούλιο προσπαθήσαμε να συμπελάβουμε και ε, ουσίες που επηρεάζουν τις αναπνευστικές οδούς. Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις για εκείνες που αφορούν το δέρμα δηλαδή το, κατηγορία τοξικότητα 3 για να το πω τεχνικά, ε, καταφέραμε να συμπεριλάβουμε τρει ουσίε ή άλλε έχουν εξερευτεί. Παρ' όλα αυτά, ήταν οι γενική έχουν εξαιρεθεί. Παρ' όλα αυτά ήταν η γενική συνένεση ότι θα προσπαθήσει να ελέγξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ποιο βαθμό στο μέλλον ε, μπορούν να συμπεριληφθούν και αυτέ οι ουσίε. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό για το Κοινοβούλιο είναι ότι ε, πέρασε η γνώμη μα στην προσαρμογή του παραρτήματος 1. Εκεί θα ακολουθηθεί η συνήθι νομοθετική διαδικασία και όχι αυτό που ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξουσιοδότηση ε, πράξης ή εφαρμοστικές πράξεις από πλευρά συμβουλίου. πράξη ε, η εφαρμοστικέ πράξει απο πλευρα συμβουλιου ευχαριστω ολους τους κοιοδη συγητέ, γιατι ειναι στεναρη η σχεση του Κοινοβουλίου απέναντι στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Καταφέραμε να περάσουμε τι θέσει μα. βελτιώσαμε αισθητά την πρόταση. Ευχαριστώ όλους ε, του συναδέλφου και κυρίω τον Γιάννο Σάντερ. Καλή τύχη στη μελλοντική του δραστηριότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον συγητή κύριο Ζέιβα. Τώρα δίνω το λόγο το λόγο έχει εξ ονόματος της Επιτροπής ο Επίτροπος κ. Τζον Νταλή. <coughs> Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Βρισκόμαστε ε, στην αρχή της πρώτης ανάγνωσης ε, για την ε, περίφημη οδηγία ΣΕΒΙΖΟ 1 και για τον έλεγχο σημαντικών κινδύνων, σημαντικών ατυχημάτων σχετικά με επικίνδυνες ουσίες. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή, τον κύριο Γιάννου Άντερ, τον οποίο εκπροσώπησε σήμερα ο κύριο Τζίμπερ, να συγχαρώ επίσης και την Επιτροπή Περιβάλλοντος περιβάλλοντος ε, και δημόσιας ασφάλειας και υγείας. Ταυμάσια η έκθεσή τους ε, και ερήμην. Θα ήθελα να συγχαρώ και τον κύριο Ράντερ για τις νέες ευθύνες που ανέλαβε, τις νέες αρμοδιότητες στην πατρίδα του. Τα βιομηχανικά ατυχήματα πολύ συχνά ε, έχουν ολέτριες συνέπειες. ή σκοτώνονται, χάνουν τη ζωή τους οι εργαζόμενοι, ε, πολλοί τραυματίζονται και υπάρχουν και ε, μακροχρόνιες επιπτώσεις. Έχουμε ρήπανση των υδάτων, πολλές εταιρείε αναγκάζονται να κλείσουν. Γνωστά βιομηχανικά ατυχήματα όπως αυτό του Σέβαζο, του Νουπάλ, της Τουλούζ, του Μπονσφίλτ. Τα ατυχήματα αυτά κόστησαν τη ζωή πολλών ανθρώπων και κόστησαν επίσης και δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή η οδηγία Σέβαζο 2 ανάγεται στο 96 και αντιμετωπίζει όλα αυτά τα προβλήματα καθορίζοντας ε, τους κανόνες για τις αρμόδιες αρχές. Κανόνες που βασίζονται στην πρόληψη ατυχημάτων μέσα από την διαχείριση της ασφάλειας, ε, της, ε, ε, των επιθέσεων επιθεωρήσεων και της χωροτακτικής ρύθμισης. Οποτεδήποτε ε, γίνονται, προκύπτουν τέτοια ατυχήματα θα πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ικανοποιημένη με το ε, συμβαστικό κείμενο ε, το οποίο καλείται να ψηφίσει το Κοινοβούλιο και το οποίο συνδέει την οδηγία με νέους κανόνες για την ταξινόμηση των χημικών ουσιών, βελτιώνει σημαντικά τους κανόνες για την πρόληψη και τον έλεγχο των ατυχημάτων. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Πρώτα απ' όλα οι κανόνες για τους ελέγχους είναι πολύ πιο λεπτομερείς και αποτελεσματικότεροι από ό,τι κατά το παρελθόν. Περιλαμβάνουν, επιβάλλουν προγράμματα για όλες τις εγκαταστάσεις και διασφαλίζουν και τη συνέχεια από τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Δεύτερον, τα δικαιώματα των πολιτών την χάνουν καλύτερων εγγύσεων. Οι πολίτες θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε καλύτερη ενημέρωση και στις επιθεωρήσεις κατόπιν τούτου η δική του συμμετοχή σε ε, χωροτακτικά προγράμματα ε, θα υπάρχει εγγύηση για τη συμμετοχή τους. Όσον αφορά τα δικαιώματα αυτά, αν δεν την χάνουν σεβασμού, τώρα οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να καταφύγουν στο δικαστήριο ε, και να επικαλεστούν τη Σύμβαση Άρχους. Είμαι πεπισμένος ότι αυτό θα επιτρέψει στους πολίτες να ασκήσουν σημαντική πίεση στους ε, αρμόδιους έτσι ώστε να τους καλέσουν να εφαρμόσουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο την οδηγία Σέβεζο, τον κανονισμό, το σχετικό. Ε, το πλαίσιο ήταν ένα σημαντικό θέμα στις διαπραγματεύσεις και τώρα επιβεβαιώνουμε το επίπεδο προστασίας των πολιτών και του περιβάλλοντος καθότι τώρα οι κανόνες θα ισχύουν και σε εγκαταστάσεις που χειρίζονται ε, ε, ουσίες ε, με τοξικότητα, κάτι που το κατά παρελθόν δεν ίσχυε. Παρόλα όλα αυτά θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να αποκτήσουμε περισσότερες γνώσεις για ουσίες ε, που επιδεικνύουν δερματική τοξικότητα. Γι' αυτό λοιπόν η Κομισιόν κάνει την εξή δήλωση. Τονίζει την πρόθεσή της να αναλύσει περαιτέρω τις, τα ατυχήματα με τέτοιου ουσίες. Η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι η σημαστική πρόταση που επιτέχθηκε σχετικά με τη δική της ε, πρόταση για την ανθρώπινη ασφάλεια και για την προστασία του περιβάλλοντος είναι καλύτερη από αυτήν που υπήρχε κατά το παρελθόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να προβεί σε εντελεχέστερη μελέτη των πιθανοτήτων και των κινδύνων ε, που μπορούν να απορρεύσουν από επικίνδυνες ουσίες που ε, χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα τοξικές. Ανάλογα με το αποτέλεσμα των αναλύσεων, η το Κομισιόν θα υποβάλει μια νομοθετική πρόταση όπου θα περιλαμβάνεται και αυτή η κατηγορία, η κατηγορία της οξίας τοξικότητας ε, στην οδηγία. Στόχος είναι να τροποποιηθεί αυξηθεί το περιθώριο εάν κριθεί απαραίτητο. Και τελειώνοντας κύριε Πρόεδρε θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει το συμβαστικό πακέτο έτσι ώστε να επιτευχθεί συμφωνία για αυτή την οδηγία κατά την πρώτη ανάγνωση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Επίτροπε, τώρα εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας το λόγο έχει ο συνάδελφος κύριος Ζακί Ενάν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό θέλαμε. Ε, μια απλή ε, καλοπιστική προσαρμογή της πρόσωψης ή μήπω μετά από τι θεομηνίες και τα ατυχήματα που είχαμε από το 1996 να προχωρήσουμε προ περισσότερη ασφάλεια για του ανθρώπου το περιβάλλον, την κοινωνία χωρί άχρηστα εμπόδια για τη βιομηχανία. Για να φτάσουμε σε αυτό το στόχο, να προσπαθήσουμε, δέχτηκα να γίνω ο ηγητής, άκουσα μαζί με άλλου και μοιραστήκαμε απόψει και θελήσαμε να περάσουμε τροπολογίε που δεν αμφισβητούν τη βιομηχανική παραγωγή, αλλά επέτρεπαν να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια για του πολίτε και για το περιβάλλον, να δίδονται νέα δικαιώματα για εκείνους που είναι οι πρώτοι εκτιθέμενοι, οι εργαζόμενοι ε, στη χημική βιομηχανία και στις μεταφορές. Ας είμαστε ειλικρινείς, δεν μας άκουσαν πάρα πολύ. Και για άλλη μια φορά ε, επικρατεί το χρήμα ε, επί των ανθρώπων υπάρχει μεγάλο χάσμα μεταξύ των μεγάλων και ωραίων λόγων που λέμε και της καθημερινή πραγματικότητα. Αυτό ισχύει για τη χημική βιομηχανία, τα εργοστάσια, τις αποθήκε και τη μεταφορά των επικινδύνων ουσιών. Για να ξεφύγουν από τους κανόνες για το Σεβέζο, ε, μείωσαν οι εταιρείε τον αριθμό ε, ε, των ουσιών ε, ε, την παραγωγή του στην αποθήκευση και ε, τα μετέφεραν σε βιτιοφόρα που μπορεί να είναι κοντά στο σπίτι σας και να εκραγούν το βράδυ που θα κοιμάστε. Θέλουμε να είμαστε καλύτερα ενημερωμένοι, καλύτερα να προστατευόμαστε. Είναι αντιφάσεις αυτές που έχουμε. Κάθε μέρα οι εργαζόμενοι σε πιο επισφαλή θέση και δεν είναι και πάντα καλά εκπαιδευμένοι. Πώς θα κάνουμε όλα αυτά μειώνοντας τις δημόσιες δαπάνες, πώς θα αυξηθεί η ασφάλεια όταν κάποιες χώρες χρησιμοποιούν αυτή τη χαλάρωση για να κάνουν περιβαλλοντικό ντάμπινγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το λόγο έχει τώρα εξ ονόματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών η συνάδελφος κυρία Μαλγκορζάτα Χάντζλικ για 1,5 λεπτό. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Η αλλαγή στην οδηγία σε Βέζο 2 απορρέουν από την ανάγκη προσαρμογής ε, ε, στον κανονισμό και όχι επειδή αυξήθηκαν τα ατυχήματα. Συμφωνώ απολύτως ότι δεν θα πρέπει να αλλάξει το σύστημα γενικότερα σε ΒΕΖΟ 2. Ως ε, σκιώδης εισηγήτρια θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενημερώνουμε το κοινό να υπάρχει δημόσια διαβούλευση και συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων και όλα αυτά να ορίζονται με τρόπο πιο συγκεκριμένο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η ενημέρωση να είναι πλήρης και κατάλληλη. Εμείς δεν επιθυμούμε να κατακλείσουμε το κοινό με άχρηστες πληροφορίες. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μεγαλύτερη ε, σαφήνεια και ε, ενημέρωση με τρόπο κατανοητό για να έχει εμπιστοσύνη ο κόσμος στην παραγωγή αυτή αλλά να εκπαιδευτεί και πώς θα φέρεται και πώς θα αντιδράσει σε περίπτωση που έχουμε ένα σοβαρό ατύχημα. Το παράρτημα είναι, είναι επίσης σημαντικό γιατί είναι κρίσιμο προς το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Γι' αυτό οι αλλαγές στο παράρτημα 1 θα πρέπει να γίνουν ε, με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία και συμφωνώ εδώ με τον κύριο Σέμπερ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Τώρα είναι η σειρά των ομιλητών εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων και εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Χριστιανοδημοκρατών. Δημοκρατών. Το λόγο έχει η συνάδελφος κυρία Σοφία Μάζεϊ Κούκοβιτς για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμο κύριε Επίτροπε, εγώ ποτέ δεν θα ξεχάσω όταν είδα τα νεκρά ε, ε, ψάρια σε ένα ποτάμι μετά από μια πυρκαγιά και διαρροή επικινδύνων ουσιών. Με φρίκη αντίκρισε αυτό το θέαμα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Έχουμε σήμερα την απαραίτητη γνώση ε, να αποτρέπουμε τέτοια ατυχήματα με τεχνολογία. Η ασφάλεια υποστηρίζεται και από πολύ υψηλέ τεχνολογίες και από ενημέρωση. Γνωρίζουμε όλε τις δυνατότητες που έχουμε, πώς μπορούμε να αποτρέψουμε αυτά τα ατυχήματα, τα ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι. Γι' αυτό ε, την έκθεση και συγχαίρω τον εισηγητή. Ίσως θα ήταν σκόπιμο να δούμε και τις επιπτώσεις ε, των ατυχημάτων αυτών στην υγεία των ζώων. Μέχρι τώρα δεν έχει ε, ε, μελετηθεί αρκετά αυτό. Θα πρέπει να ενημερώνουμε για την πρόληψη και για την αντίδραση σε περίπτωση ατυχημάτων. Η εισπνοή ατμών και αεροζόλ που περιέχουν επικίνδυνα σωματίδια είναι κάτι που δεν το αντιλαμβανόμαστε πάντα εκ πρώτης όψεως. Είναι πολύ σημαντικό και την υγεία μας την αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική είναι όταν τη χάνουμε. Όταν ο οργανισμός μας παθαίνει βλάβες. Ευχαριστώ. Στο όνομα της ομάδας Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το λόγο έχει η συνάδελφος κυρία Όσα Βέστλουντ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Άντερε και τον Επίτροπο Νταλή, καθώς και τους, ε, τη Γανική Προεδρία και όλους τους ε, υπολείπους εκπροσώπους ε, των πολιτικών ομάδων για την ε, καλή συνεργασία που είχαμε. Για τη δική μου πολιτική ομάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ύψιστη προστασία της δημόσιας υγείας μέσω αυτής της οδηγίας και νομίζω ότι επιτύχαμε ναι, να εκπληρώσουμε αυτή μας τη φιλοδοξία. όλα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής πρόληψης των μεγάλων ε, ατυχημάτων που εντάσσεται με τη σειρά του στο πλαίσιο της ε, ε, της μεγαλύτερης ασφάλειας για την αντιμετώπιση τέτοιων μεγάλων κινδύνων από πλευρά των κρατών μελών. Ενισχύεται λοιπόν η δράση μας, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια. Τα κράτη-μέλη πρέπει να διεξάγουν επιθεωρήσεις. Υπάρχουν πιο μεγάλοι περιορισμοί στις συνέχεια αναφερόμαστε στο αποτέλεσμα ντόμινο για να αποφύγουμε ακόμη μεγαλύτερα ατυχήματα. Εξασφαλίζουμε καλύτερη ενημέρωση τη κοινή γνώμη. Επίση, εξασφαλίζουμε ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλε τι πληροφορίε ε, για όλε τι ουσίε ε, και την ταξινόμησή του και τι διάφορε νέε κατηγορίε. Αλλά πέρα από την προστασία του περιβάλλοντο και των ανθρώπων, ε, διευρύνουμε επίση το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία, ούτω ώστε να είναι καλύτερη η ενημέρωση τη κοινή γνώμη. τώρα, θεωρώ θεωρώ ότι θα πρέπει να τροποποιηθούν ε, αυτά τα κριτήρια όπως και κάνουμε μέσω αυτού του βασικού νομοθετήματος ε, σχετικά με τις ε, πράξεις κατεξουσιοδότηση πιστεύω ότι είναι η μόνη λύση που πρέπει να δεχθούν τα κράτη-μέλη ουδάλλως δεν θα επιτύχουμε το στόχο μας και ελπίζω να έχουμε καλή έκβαση ψηφοφορίας αύριο το πρωί ευχαριστώ Εξ ονόματος της Συμμαχίας και Δημοκρατών για την Ευρώπη το λόγο έχει ο συνάδελφος κύριος Βλάτκο Τόντοροφ Παναγιώτοφ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, χρειαστήκαμε πάρα πολύ χρόνο για να καταφέρουμε να συμφωνήσουμε για την οδηγία σε ΒΕΣΟ 3, νομίζω ότι τώρα μπορούμε να δηλώσουμε ικανοποιημένοι με τα εκτευθέντα αποτελέσματα, τα μεγάλα ατυχήματα στο Νεπάλ, στην Ινδία, το 1984, το 2001 στην Τουλούζη και άλλα μας έδειξαν ότι οφείλουμε να αναθεωρήσουμε την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία στον τομέα αυτό. Το Συμβούλιο δεν ε, ε, ήταν τόσο φιλόδοξο όσο το Κοινοβούλιο, κυρίως ε, ως προς την πρόσβαση του κοινού στις τεχνικές αυτές πληροφορίες. Καταφέραμε πάντως να επιβάλλουμε την άποψή μας και όχι μόνο αυτό, αλλά καταφέραμε Κάποιε ουσίε να μην υπάγονται στι πράξει ε, ε, κάτι εξουσιοδότηση, αλλά να περνούν από τη συνήθη νομική, ε, ε νομοθετική διαδικασία. Διευρύνεται ε, μέσα από την έκθεση, μέσα από την νέα πρόταση μάλλον, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας Παρότι εγώ λυπάμαι, διότι δεν ήμασταν υπαρκώ φιλόδοξοι για την πρόσβαση στις πληροφορίες και τον κατάλογο των επιχειρήσεων που εμπορεύονται αυτές τις ουσίες. Πλην όμω, δηλώνουμε ικανοποιημένοι διότι έχουμε νέους κανόνες για την προστασία, για την διαφάνεια, για την πρόσβαση στις πληροφορίες για τους πολίτες. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο που εργάστηκε τόσο σκληρά για αυτό το θέμα. Ε, ακολουθεί στο βήμα εξ ονόμου της ομάδας των Πρασίνων της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας ο συνάδελφος κ. Κάρλ Σλίτερ για ένα λεπτό. Eh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον Γιάννου Σαντέρ ε, και να τον συγχαρώ για τα όσα συνέβησαν στην Ουγγαρία. Ε, μετά από πολύ δύσκολες ε, διαπραγματεύσεις ε, όπου αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες λόγω της αναταξινόμησης των ουσιών διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε μεγαλύτερη προστασία στις μονάδες παρά τη νέα ταξινόμηση. Εάν θέλουμε λοιπόν να προστατεύσουμε την υγεία και να αποφύγουμε τα ατυχήματα δεν έχουμε επιτύχει το στόχο μας και τελικά καταλήξαμε σε μια συμφωνία που εντάξει λειτουργεί καλύτερα σε σχέση σχέση με την προηγούμενη οδηγία σε ΒΕΣΟ είναι πάρα πολύ σημαντικό που δεν επέβαλε το Συμβούλιο τις αρχικές κατηγορίες ε, ουσιών που είχε ε, προτείνει. Θα ήθελα να διερευνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσα σας είπα για περί ασφάλειας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν γίνεται το κόστος ε, να έχει μεγαλύτερη να είναι τόσο επαχθές ούτως ώστε να μην τα καταφέρνουν οι επιχειρήσεις και τελικά να μην συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις. Δεν πρέπει να βαρύνει αυτό αυτό τους φορολογουμένους. Της ομάδος των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών το λόγο έχει η συνάδελφος κυρία Άννα Ρόσμπακ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζουν κοντά σε ε, βιομηχανίες, που, εταιρείες που εργάζονται με επικίνδυνες χημικές ουσίες. Άρα απειλείται η ζωή τους, η υγεία τους, αλλά και το περιβάλλον. Από τον Ιούνιο του 2015... Ε, οι 10.000 αυτές εταιρείες θα έχουν πιο αυστηρούς κανόνες να πληρούν για να αποτρέπονται τέτοια ατυχήματα με επικίνδυνες τοξικές ουσίες και να ενημερώνονται οι πολίτες. Θετικά είναι όλα αυτά. Αλλά επειδή γνώρισε μεγάλη αντίσταση στο Συμβούλιο, η πρόταση και η κατάσταση για τους ε, πολίτες και για το περιβάλλον δεν είναι καθόλου ιδανική. Θα πρέπει συνεχώς να εξασφαλίζεται η προστασία και ασφάλεια των πολιτών που ε, κατοικούν κοντά σε τέτοιες επιχειρήσεις. Το πιο θετικό από όλα είναι ότι βελτιώνεται τώρα η ενημέρωση των πολιτών της Ένωσης. Δεν θα πρέπει μόνο να ε, έχουμε πρόληψη αλλά και ενημέρωση και μέσω του διαδικτύου και αυτό υποστηρίζω την πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, για την Ευρώπη της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας δίνω τώρα το λόγο στον συνάδελφο κύριο Ρέστε Ρώση για ένα λεπτό. Συμφωνούμε με τον εισηγητή ότι το πρώτο και δεύτερο τμήμα του παραρτήματος ε, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με κατεξουσιοδότηση πράξης. Ε, πρέπει να πούμε ότι το πεδίο εφαρμογή ε, δεν ε, είναι ισορροπημένο και θα οδηγήσει ε, σε αύξηση του βάρους που δεν είναι σε σωστή αναλογία με τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Πέρα από αυτό, μια σημαντική αύξηση του διοικητικού κόστους, αυτό θα οφείλεται στο ότι είναι απαραίτητο αυτός ο οργανισμός, ο CLP, να ε, προσαρμοστεί στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από τους βιομηχάνους που ζητούν εφαρμόζεται το B-Plan, ε, δηλαδή το πρόγραμμα αυτό είναι πολύ καλά παγιωμένο και έχει αποδειχτεί ότι λειτουργεί σωστά. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, το ευρύ πεδίο εφαρμογής, έχουμε αποδείξει ότι κυρίως οι ρυθμίσεις αφορούν τη βιομηχανία. Εμείς ε, δεν ε, θεωρούμε ότι αυτός είναι σωστός ε, τρόπος για να νομοθετούμε, γιατί τελικά πρέπει να επικρατεί η πραγματικότητα. Να προσθέσουμε τα αντικείμενα που αφορούν τις offshore ε, πλατφόρμες ε, και τις εγκαταστάσεις για την αφαλήνωση. Της Ευρωπαϊκή Ενωτικής Αριστεράς, της Αριστεράς των πρασίων των Βορείων Χωρών, η συνάδελφος κυρία Άλντα Σούσα. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, οι επικίνδυνε ε, ουσίε ε, και οι επιπτώσει που έχουν στη βιομηχανία είναι μια δυσάρεστη αλήθεια της σημερινής οικονομίας. Τώρα, είναι αναγκαίο, δεν είναι μόνο δικαίωμα να μπορούν οι πολίτες να συμμετάσχουν στη λήψη αποφάσεων για να περιορίσουμε τις ζημιές και να μπορέσει η κοινωνία των πολιτών να προστατευτεί από αυτέ τι καταχρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν σε πρώτη προτεραιότητα να αντιμετωπίσουμε τι τις συνέπειες της χρήσης αυτών των ε, ουσιών, ε, αλλά όχι μόνο. Ε, οι φτωχότεροι των φτωχότερων στην Ουγγαρία εγκαταλείφθηκαν. Βλέπουμε επίσης τι συνέβη στην Ινδία, στον Νεπάλ, εκατοντάδες χιλιάδες θύματα εγκαταλείφθηκαν στην τύχη τους όταν οι επιχειρήσεις συνέχισαν ανενόχλητες τη δράση τους. Δεν μπορούμε στην Ευρώπη να το ξεχάσουμε αυτό. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, μεγαλύτερη διαφάνεια και να σταματήσουμε τη δράση αυτών των εταιριών. Δεν βλέπω στην αίθουσα τον συνάδελφο κύριο Φραντς Ομπεμάια και περνούμε στους άλλους εγγεγραμμένους ομιλητές. Δίνω αμέσω το λόγο στη συνάδελφο κυρία Μορκουνέιτε Μικουλιενένε για 1,5 λεπτό aplinkos apsaugos politikos raida dažnai dėja yra tokia kad paprastai nauji Κοιτάξτε, η προστασία του περιβάλλοντος κατ' ουσίαν απαιτεί νέες ρυθμίσεις όταν προκύπτουν μεγάλα ατυχήματα. Ο στόχος της νομοθεσίας δεν είναι μόνο να ανταποκρινόμεθα, να αντιμετωπίζουμε, αλλά και να προλαμβάνουμε τέτοιου είδους ατυχήματα. Στο μέλλον ε, θα πρέπει να τονίσουμε περισσότερο την πρόληψη. Και σήμερα η οδηγία που συζητάμε έχει ακριβώς αυτό ως στόχο. Θέλουμε να συνδυάσουμε τις νομικές απαιτήσει με την τεχνολογική πρόοδο. Πρέπει όμως να πούμε ότι απλά προσπαθούμε να προλάβουμε την πραγματικότητα. Παραδείγματο χάρη οι τεχνικές, κάποιες τεχνικές αλίευσης σε ανοιχτή θάλασσα δεν εμπίπτουν στο πεδίο της εφαρμογής ανάλογα με το πώς κινείται το σκάφος και όταν ε, προκύπτει το ατύχημα οι συνέπειες εξακολουθούν είναι πολύ σημαντικές. Ε, είναι λοιπόν σημαντικό ε, το ότι υπάρχει αυτή η οδηγία και πιστεύω ότι η κοινωνία πρέπει να έχει την ε, δυνατότητα να συμμετέχει στη λήψη των αποφάσεων γιατί όλα αυτά ε, θα συμβάλλουν στο να υπάρχει καλύτερη περιβαλλοντική προστασία. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι η κοινωνία θα έχει πρόσβαση στην ε, ενημέρωση, πρόσβαση στους ελέγχους. Και θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Είναι ο συνάδελφος Ματίας για λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σέβεζο, Ενσεντέ, τουλούς ε, τα ονόματα αυτά είναι ονόματα πόλεων για πολύ μεγάλα ατυχήματα όπου όχι μόνο υπήρξε περιβαλλοντική καταστροφή αλλά και θύματα καταστροφή ιδιωτικής περιουσίας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε οι κίνδυνοι αλλά και η πιθανότητα να επαναληφθούν τέτοιου είδους ατυχήματα να περιοριστούν. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό πρώτον με το να γίνονται έκτακτες επιθεωρήσεις να μην είναι αυτό ρουτίνα και οι άνθρωποι που ζουν κοντά σε αυτές τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις να είναι πολύ καλά ενημερωμένοι για το τι ακριβώς συμβαίνει και στην, σε κάποια σοβαρή περίπτωση να ε, διαδίδεται ταχύτατα η πληροφορία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορούν να σωθούν ανθρώπινες ζωές με τον τρόπο αυτό. Πιστεύω λοιπόν ότι το ε, Συμβούλιο εδώ ε, δεν ε, έδειξε τη δέουσα προσοχή. Παρεπιπτόνως λείπουν εδώ οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου. Ε, ίσως να υπάρχουν κάτι να υπάρχουν πράγματα πιο σημαντικά, αλλά θα ήταν καλό να μας εξηγήσει το Συμβούλιο γιατί νοθεύτηκε η νομοθεσία. Αυτό θα μου άρεσε να το ακούσω. Πάντως, ε, ισχυρή νομοθεσία προκαλεί και εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη στο να εφαρμόζονται οποτεδήποτε συζητώνται τα ε, μεγάλα προγράμματα στις, στα κράτη-μέλη γιατί οι πολίτες έχουν πάντα επιφυλάξεις και νομίζω ότι προκαλεί εμπιστοσύνη και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και με το να συνδέονται καλύτερα οι υπηρεσίες, καλύτερη λοιπόν συνεργασία και επικοινωνία και επουδενή όποτε υπάρχουν ε, επαφή με τέτοιου είδους ε, μεγάλες εγκαταστάσεις να μην αντιμετωπίσετε αυτό ε, στο πλαίσιο μιας ρουτίνας. Πολύ ωραία. Το λόγο έχει ο κύριος Γκέρλινγκ, η κυρία Γκέρλινγκ, με συγχωρείτε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βεβαίω όλοι υποστηρίζουμε ενεργά την πρόληψη σοβαρών ατυχημάτων που αφορούν ε, ποσότητες ε, επικινδύνων ουσιών. Γνωρίζω ότι δεν ήταν εύκολο αυτό το θέμα για να ικανοποιήσει όλους. Ήταν πολύ έντονη η συζήτηση για το πεδίο εφαρμογή και τη δυναμική βάση για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την ενημέρωση των πολιτών. Γι' αυτό χαίρομαι πολύ που έχω την ευκαιρία να συγχαρώ την ομάδα που το χειρίστηκε με υπομονή και επιμονή. Είναι πολύ ε, πρόσδεκτη η νέα πρόταση. Ξέρω ότι το νέο πακέτο σε θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τους κανονισμούς CLP για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία. Ε, γνωρίζω ότι υπήρχε πρόβλημα και ε, επίσης υπήρχε και πρόβλημα επικαλύψεων που πιστεύω ότι τώρα αποφεύγει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Επίτροπο για τη σημερινή του πρόσθετη δήλωση η επιθεώρηση και η ανάλυση σε πραγματικό χρόνο είναι πολύ σημαντικό γιατί έτσι βελτιώνεται και η πολιτική και η νομοθεσία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η οδηγία σε Βέζο 2 είναι ένα απαραίτητο βήμα για την πρόληψη τέτοιων ατυχημάτων όπως είδαμε στην Τουλούζη ε, για παράδειγμα, στο Σεβέζο και αλλού και είχαμε πολλές και υλικές ζημιές και περιβαλλοντικές ζημιές ε, και μεγάλο κόστος. Η οδηγία αυτή είναι σημαντική διότι επιβάλλει στα κράτη-μέλη και τις εταιρείες ε, ε, κάποιους κανόνες για να προλαμβάνονται τα ατυχήματα και να περιορίζονται οι συνέπειες τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει συστηματικά να κάνει τέτοιους κανονισμούς και μάλιστα πιο αυστηρούς. Η αναθεώρηση της οδηγίας αυτής θα βελτιώσει ε, το συντονισμό με τον εμφιστάμενο κανονισμό και θα σταματήσει τους διπλούς ελέγχους και τη διπλή νομοθεσία. Ιδιαίτερη επιθεωρήσεις θα πρέπει να αφορούν και τους υπεργολάβους, διότι πολύ συχνά αυτοί είναι οι πέτοι και δεν ε, συμμορφώνονται με την νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκπροσωπεί τους πολίτες της Ένωσης θα πρέπει να συμμετέχει πλήρως στις συζητήσεις. Γι' αυτό συμφωνώ με τον εισηγητή ότι οι αλλαγές στον παρόντο κανονισμό πρέπει να γίνουν μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Να συμμετέχει το Κοινοβούλιο και να ενημερώνεται και από την Επιτροπή σε τακτά χρονικά διαστήματα για τέτοιου είδους ατυχήματα και πώς εμεί ε, απαντούμε και αντιδρούμε σε αυτά. Ο κόσμος θα πρέπει να έχει εύκολη πρόσβαση ε, σε αξιόπιστη ενημέρωση για τις απειλές και για τον τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση που γίνει ένα τύχημα. Το διαδίκτυο είναι ένα καλό εργαλείο που θα πρέπει να χρησιμοποιείται το συντομότερο, να αρχίσει ενημερωτική εκστρατεία για τη νέα ταξινόμηση τοξικότητα ουσιών και απειλές για τη ζωή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Μέρκης για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επίτροπε, πριν από 12 χρόνια στο NCDS στην Ολλανδία ε, θυμάστε ε, την έκρηξη σε ένα εργοστάσιο ε, πυροτεχνημάτων έκανε το γύρο του κόσμου η ε, είδηση 22 νεκρούς στην περιοχή στο Μόρδαϊκ θυμάστε ε, ήταν γνωστό τι συνέβαινε στην εταιρεία αυτή ε, αλλά τους είχαν δώσει μεγάλο περιθώριο ελιγμών. Κάθε φορά που γίνονται τέτοια ατυχήματα, απαντάμε με τον νόμο. Αλλά εντάξει ο νόμος, θα πρέπει να γίνεται και η σωστή εφαρμογή του νόμου. Τα ξέραν όλα αυτά και στο έσχεται. Είναι καλή η οδηγία αυτή και η αναθεώρηση γιατί αυξάνεται πολύ η διαφάνεια για τους πολίτες, η ενημέρωση και δημιουργείται έτσι εμπιστοσύνη και κυρίω το γεγονό ότι όλα αυτά είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι πολύ εύκολο οι πολίτε να ενημερώνονται. Παραμένει όμως ένα πρόβλημα με την ενημέρωση. η ε, τοπική αυτοδιοίκηση, η αρμόδια αρχή, εν περιπτώσει, δεν έχει πάντα την πραγματογνωμοσύνη για να κάνει αυτές τις επιθεωρήσεις. Θα πρέπει να γίνονται με σωστό τρόπο και οι έλεγχοι και να ενημερώνονται και οι υπηρεσίες που παρέχουν τις πρώτες βοήθειες και πρέπει να αντιδράσουν για να δημιουργεί και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη της πολίτες. Ευχαριστώ. Ο κύριο Αρσένη, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Τα... Συντάμε μια πάρα πολύ σημαντική οδηγία. Τα ατυχήματα με επικίνδυνε ουσίες συμβαίνουν σπάνια. Συμβαίνουν όμως, όταν συμβαίνουν όμω οι επιπτώσει είναι τραγικέ. Τραγικέ για του πολίτε, τη περιοχή, είναι μακροχρόνιε και κρατούν πολλέ γενιές. Καταφέραμε να βελτιώσουμε την νομοθεσία όμως υπάρχουν θέματα για τα οποία δεν τολμήσαμε. Δεν τολμήσαμε να συμπεριλάβουμε παραδείγματος χάρη τις εξέδρες εξόρυξης πετρελαίου. Παρά την τραγική εμπειρία σε πολλές χώρες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά την τραγική εμπειρία του ατυχήματος στο Μεξικό και παρά τις τραγικές επιπτώσεις και για την οικονομία και για τη θαλάσσια ζωή και τους πολίτες. Θεωρώ ότι πολλές φορές οι πολίτες περιμένουν περισσότερα από εμάς, από όλους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και πραγματικά εύχομαι τις επόμενες φορές να συμπεριλάβουμε τις εξέδρες και να είμαστε πιο συνεπείς στα αιτήματα των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα λοιπόν ε, θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία Catch DI. Ξεκινάμε με ε, την κυρία Κάντενμπαχ. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε, ως Αυστριακοί εμείς ε, το 2010 από την καταστροφή στην Ουγγαρία ε, πληγήκαμε οι πολίτες ανησύχησαν πάρα πολύ, η ανασφάλεια ήταν πολύ μεγάλη και γι' αυτό λοιπόν χαιρετίζω αυτή την πρόθεση, το ΣΕΒΙΖΟ 3, ακόμα ε, και αν συμφωνώ με τον κύριο Γκρότε ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη υπήρξε προσπάθεια ε, χαλάρωσης. Ε, εγώ θεωρώ ότι χρειαζόμαστε τη διαφάνεια, την ενημέρωση και αυτό που χρειαζόμαστε κυρίως είναι η οικονομική εξασφάλιση, γιατί δεν είναι δυνατόν ε, το κόστος ε, να μετακυλίεται στους πολίτες. Εγώ λοιπόν σας παρακαλώ θερμά να υπάρχουν προγράμματα έκτακτης ανάγκης που να συμπεριλαμβάνουν τους πολίτες ε, που πραγματικά να λαμβάνουν υπόψη τους τις ανησυχίες των πολιτών. Καταλήγω, όλα είναι χημεία, αλλά η επικίνδυνη χημεία πρέπει να ελέγχεται και το ΣΕΒΕΖΟ 3 θα μας προσέφερε τη δυνατότητα να είμαστε ακόμα πιο αυστηροί. Πολύ ωραία το λόγο. Ε... Κυρία Ριβαζή, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους ε, όλος ιδιαίτερα τον κύριο Άντερ και τον κύριο Σέμπερ για το έργο τους σε αυτή την έκθεση. Είναι γεγονός ότι η οδηγία του Σεβέζο και το ατύχημα της Τουλούζης Άζεντεφ, θυμάστε, 21 Σεπτεμβρίου του 2011 Νητρικό αμμόνιο εξεράγει δεξαμενή 31 νεκροί, 2.500 ε, ε, τραυματίες, τρομερές ζημιές και ακόμα περισσότερες ε, και σήμερα παραμένουν οι συνέπειες. Ε, το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν οι υπεργολαβίες ε, που οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν ενήμεροι, δεν ήταν ε, σωστά κατερτισμένοι. Χαίρομαι, εν περιπτώσει, για το τελικό αποτέλεσμα, για τη διαχείριση βιομηχανικών κινδύνων. Θα πρέπει να ενημερώσουμε τους πολίτες, γιατί οι εταιρείε κάνουν οικονομία στην ασφάλεια. Υπάρχει σύμβαση του άρχους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ενημέρωση του κοινού, των πολιτών, για τη διαφάνεια και εκ των όνων για να έχουμε ένα σχέδιο διαχείρισης αποτελεσματικό. Ένα ίσως αρνητικό Επίτροπε, το μόνο δεν υπάρχει αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων των σοβαρών ατυχημάτων και πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα επιχειρήσεις. Γι' αυτό είναι έλλειψη ε, σε αυτή την οδηγία, πρέπει να καλυφθεί. Πάσκα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε, η θέση σε ισχύ του κανονισμού 1272 του 2008 ήταν το κίνητρο για την προσαρμογή της οδηγίας Σέβεζο 2. Αυτή η προσαρμοσμένη οδηγία οδηγεί σε ένα καλύτερο σύστημα ταξινόμησης ε, των χημικών ουσιών. Και πλέον έχουμε τρεις ε, κατηγορίες τοξικών ουσιών και παράλληλα υπάρχουν και πέντε ε, διαφορετικές κατηγορίες έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες. Παρ' όλα αυτά λείπουν κάποια στοιχεία ασφάλειας. Λείπει κυρίως η ρύθμιση των υπεργολαβών ε, Επίσης ε, λείπει και ένας ε, κανονισμός για την αποθήκευση των επικίνδυνων ουσιών σε εγκαταστάσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Ένα άλλο μειονέκτημα της οδηγίας είναι ότι τα κρατημέλη είναι σε θέση να προβλέπουν εξαιρέσεις. Ε, πολλές καταστάσεις τους προηγούμενης χρονιάς μας ε, έδειξαν ότι εκτός από τους τεχνολογικούς κινδύνους πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και τους φυσικούς κινδύνους. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να στηρίξουμε όλες τις ε, τροπολογίες της Επιτροπής Ήτρε που ε, προσπαθεί να εξαλείψει τα προβλήματα που υπάρχουν από την πρόταση της Επιτροπής. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Επίτροπος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη πρέπει να σας πω ότι τελικά καταλαβαίνω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε στην δέσμη μέτρων που θα ψηφιστούν αύριο. Αυτή η δέσμη μέτρων θα επιτρέψει στα κρατη να εξασφαλίσουν καλύτερη εφαρμογή των πολιτικών τους για την πρόληψη και τον έλεγχο πολιτικών ε, σχετικά με μεγάλα ατυχήματα και επικίνδυνες ουσίες. Αυτές οι ουσίες ορίζονται τώρα πλέον ε, στη νέα ταξινόμηση και συμμορφίζουν πλήρως με τη νέα ταξινόμηση. Η Επιτροπή είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Εγώ θα ενημερώσω τους ε, συναδέλφους μου, τον κύριο Ποτόκνητς, ε, κυρίως για το αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς, λέει η Επίτροπος και τώρα το λόγο έχει ο εισηγητής κύριος Ζέμπα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι η συζήτηση κατέδειξε με απόλυτη σαφήνεια ότι δεν είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς με αυτό το συμβασμό, αλλά έτσι είναι οι συμβασμοί. Θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε περισσότερο, αλλά εδώ μας μπλοκάρισε κυρίως ε, το Συμβούλιο. Εξάλλου η συζήτηση κατέδειξε με σαφήνεια ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στη σωστή εφαρμογή. Αυτό είναι βασικό πρόβλημα. Ε, ορισμένα κρατημέλη. Δυστυχώς είναι πολύ χαλαρά στην εφαρμογή. Νομίζω λοιπόν ότι ειδικά εδώ στο ε, ΣΕΒΕΖΟ 3 πρέπει να αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία γιατί πρόκειται για ανθρώπινες ζωές που βρίσκονται σε κίνδυνο αν οι άνθρωποι αυτοί ζουν κοντά σε χημικές εγκαταστάσεις. Ε, πρέπει ε, τους κινδύνους να τους διαχειρίζεται κανείς σωστά. Εξάλλου κατέστη απόλυτα σαφέ ότι τα εργαλεία που υπάρχουν όπως τα προγράμματα έκτακτης ανάγκης αυτά θα πρέπει να είναι σαφή, να περιλαμβάνουν την κοινή γνώμη, έτσι ώστε οι πολίτες ε, να γνωρίζουν αν συμβεί ένα τύχημα πώς πρέπει να αντιδράσουν. Νομίζω λοιπόν με καλή επεξεργασία αυτών των προγραμμάτων μπορούμε να σώσουμε πάρα πολλές ε, ζωές. Αυτό είναι καθοριστική σημασία. Σημαντικό είναι να εκπαιδεύονται σωστά και οι φύλακες ε, που βρίσκονται μέσα σε μια εγκατάσταση. Είναι σημαντικό σημαντικό οι πολίτες να νιώθουν εμπιστοσύνη και κυρίως να υπάρχει πρόληψη και όσον αφορά την πρόληψη ε, καθοριστική σημασίας είναι ε, και η διαχείριση επιτόπου. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να θεωρούμε ότι είμαστε ευτυχείς ε, ε, κυρίως για το ότι ε, το Κοινοβούλιο συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα 1. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην μας παραγωνίσουν. Νομίζω ότι αυτό το καταφέραμε και γι' αυτό λοιπόν τελειώνοντας θέλω να πω ότι η συμβαστική πρόταση σε γενικές γραμμές είναι καλή. Θα θέλαμε να προχωρήσουμε παραπάνω, αλλά στο πλαίσιο μια συμφωνίας με το Συμβούλιο και την Κομισιόν νομίζω ότι μπορούμε και εμείς να συμφωνήσουμε. Κύριε Σίμπα, δέχεστε μπλε κάρτα, παρακαλώ. Κοιτάξτε, μπλε κάρτα, γιατί ακούσαμε πάρα πολλές ε, επικριτικές φωνές. Ξέρω ότι συνάδελφος κύριος ε, Ζήμπα γνωρίζει πολύ καλά τη διαδικασία στο Κοινοβούλιο και υιοθέτησε την έκθεση του κυρίου Άντερ. Και ερωτώ, ε, τι θα γίνει τώρα στην πρώτη ανάγνωση όπου ε, το 65% αφορά θέματα περιβάλλοντος και ερωτώ τον εισηγητή μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια αν ε, υπήρχε εδώ και το Συμβούλιο και αν το είχαμε πάει στη δεύτερη ανάγνωση ε, ξέρω αγαπητέ Ρίχαρτο ότι εσύ απλά αντικαθιστάς τον εισηγητή αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να έχω ακούσει την άποψη του εισηγητού επί του θέματος όπως ε, είπε και εσύ Ματίας Γκρότε, εσύ είσαι ο ε, πρόεδρος Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος ε, και υπό την αιγίδα σου δουλεύουμε σωστά. Νομίζω για αυτό το θέμα δεν θα βοηθούσε τίποτα το να υπάρχει μια δεύτερη ανάγνωση. Ε, νομίζω ήταν σωστό από, τον, από πλευράς εισηγητού να καταθέσει την έκθεση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η Κομισιόν υιοθέτησε την άποψη να εξετάσει τακτά χρονικά διαστήματα ποιες ουσίες ε, πρέπει να προστίθενται. Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο κύριος ε, Ποτότσνικ για να ασκήσει πίεση και να έρθει πιο πολύ κοντά στις δικές μας απόψεις. Ευχαριστούμε. Έκλεισε λοιπόν η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12. Τώρα, περνάμε στην δήλωση της Αντιπροέδρου ε, της ε, Επιτροπής ε, σχετικά με το γενετικό ακροτηριασμό εκ μέρους λοιπόν της κυρίας Άστον. Θα λάβει το λόγο Επίτροπος κύριος Ντάλι, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάθε είδους βίας με βάση το φύλλο ε, συνιστά απαράδεκτη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων